Possiamo iniziare? Λοιπόν, ξεκινάμε. Περνάμε στο 11. Αφού χαιρετήσω τους επισκέπτες μας, που είναι παρόντες στην Επιτροπή Γεωργίας, Έχουμε επίσης και τους φιλοξενούμενους της κυρίας Πάουλσον και Ρόντοστ. Σας καλωσορίζω όλους. Ξεκινάμε λοιπόν τη σημαντική αυτή νομίζω ακρόαση για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας αυγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συζητήσουμε λοιπόν για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο τομέας αυτός. Θα κάνουμε μια αξιολόγηση εταιρικών παραγόντων που επηρεάζουν την αγορά των αυγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μιλήσουμε για τις εμπειρίες των ομιλητών και για τις μελλοντικές προοπτικές. Καλωσορίζω τρεις εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα πάρουν το λόγο. Μετά από τις παρουσιάσεις τους θα υπάρξει νομίζω χρόνος για ε, ερωτήσεις και απαντήσεις ανάμεσα στους συναδέλφους που θέλουν να πάρουν μέρος. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Μάρκ Williams, Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εμπορίου Χονδρικής Αυγών και Πουλερικών. Θα μας μιλήσει για την ανταγωνιστικότητα της, βιομίας, της βιομηχανίας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της απελευθέρωσης της αγοράς. Μετά θα ακούσουμε τον Μίχελ Γιούσε που είναι υπεύθυνο της ε, αυστριακής βιομηχανίας και οικονομικής δραστηριότητας γύρω από τα πουλερικά που θα μας μιλήσει για τις προσδοκίες των καταναλωτών και θα κλείσω με τον κύριο ε, Νιεβιαντόμσκι, διευθυντή της εταιρείας Φάρμιο πολωνικής εταιρείας που θα μας μιλήσει για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας που ασχολείται με τα πουλερικά και τα αυγά. Ξεκινάω δίδοντας το ρόλο στον κύριο Williams. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να μείνουμε σε μισή ώρα και για τους τρεις, γύρω στα δέκα λεπτά πάνω κάτω για τον καθένα σας. Ο κύριος Williams έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλου. Σα ευχαριστώ που μου δίνετε δυνατότητα να μιλήσω εδώ στην Επιτροπή σα σήμερα. Θα ήθελα να σα ενημερώσω για τα όσα ε, εμεί θεωρούμε εύλογε ανησυχίε και σημεία προβληματισμού σε ό,τι φορά τι μελλοντικέ εμπορικέ διαπραγματεύσει και συμφωνίε. Χωρί επιπλέον καθυστέρηση λοιπόν μπορώ να προχωρήσω. Ποιοι είμαστε εμεί, Η UWeb είναι Ευρωπαϊκό Σωματείο που εκπροσωπεί τα συμφέροντα της ε, βιομηχανίας ε, αυγών σε όλους τους τομείς ε, μεταποίησης, συσκευασίας και εμπορίας. Εμείς δηλαδή παίρνουμε τα αυγά και τα φέρνουμε στην αγορά. Η βιομηχανία αυγού θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα επιτυχής είχαμε μόνο ένα ε, light, ε, ελαφρύ καθεστώς ε, κοινής γεωργικής πολιτικής, το οποίο μας βοήθησε και μας επέτρεψε να είμαστε επιτυχείς, αποτελεσματικοί και καινοτόμοι στη δράση μας. Και βεβαίως πρέπει να αντιποκρινόμαστε στην ζήτηση των καταναλωτών. Στα καταστήματα βλέπετε όλες τις διαφορετικές μορφές αυγού που διατίθενται μας διακρίνει υψηλός βαθμός ευθύνης. Το βασικό σημείο και ε, πλεονέκτημα της βιομηχανίας μας είναι η ε, επιστηστική ασφάλεια. Υπάρχει πλήρης ανιχνευσιμότητα, υπάρχουν πολλά καθεστώτα διασφαλίσεων που λειτουργούν ε, στα κράτη-μέλη για την και η των ζώων και η προστασία του περιβάλλοντος είναι εξαιρετικά σημαντικά σημεία για μας. Θα ήθελα λοιπόν να σας επισημάνω μία έκθεση που ζήτησε ε, το LEI, Ολλανδικό ε, Ινστιτούτο. Είχαμε κάνει και μία προηγούμενη μελέτη το 2003 που επικαιροποιήθηκε το 2005. Όμως το 2011 θεωρήσαμε σημαντικό να επικαιροποιηθεί εκ νέου. Σε αυτή την έκθεση εξετάσαμε το κόστος ε, παραγωγής και μεταποίησης των αυγών σε 7 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως βλέπετε στις οθόνες σας, Πρόκειται για του ε, έξι μεγαλύτερου παραγωγού ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω η Γερμανία είναι από του μεγαλύτερου παραγωγού, αλλά επειδή είναι ιδιαίτερα παρόμοιε οι αγορέ ή ο τρόπο παραγωγή στην Ολλανδία και στη Γερμανία, χρησιμοποίησαμε μόνο την Ολλανδία και προσθέσαμε και τη Δανία. Μη κράτη-μέλη Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ουκρανία, γιατί βρίσκονται στα ανατολικά μα σύνορα, προφανώ, οι Ηνωμένε Πολιτείε, Αργεντινή και Ινδία. Επιλέξαμε αυτέ τι τρει χώρε, γιατί είναι οι τρει χώρε που εξάγουν τα περισσότερα προϊόντα αυγού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα εκπροσωπούν το 75% των εξαγωγών. Σε την νομοθεσία που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάναμε κάποιες ε, προβλέψεις το 2012, γιατί από τις αρχές του 2012 ξεκίνησε η απαγόρευση των ε, συμβατικών κλοβών. Εξετάσαμε και διάφορα σενάρια για την ε, μελλοντική ανταγωνιστική μας θέση. Για όσους γνωρίζετε, εξετάσαμε τα βασικά ε, στοιχεία που είναι ε, οι ζωοτροφές, ε, η στέγαση, ο εξοπλισμός, οι ενεργειακές δαπάνες αλλά και οι δαπάνες μεταφορών, γιατί πρέπει βεβαίως να φτάσουν στην αγορά. Εδώ σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε στην αριστερή στήλη το μέσο κόστος παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπετε ότι είμαστε πολύ παραπάνω από τις προηγούμενες ε, τέσσερις χώρες που ανέφερα. Αντίστοιχο εγχείρημα κάναμε και για το κόστος μεταποίησης ε, για την ε, σκόνη όλου του αυγουπλήρους αυγού. Δηλαδή το αυγό που το έχουμε βγάλει από το κελυφός του και το έχουμε αποξηράνει. Το κόστος εδώ είναι πολύ ε, ε κοντά σε, στο κόστος των ΗΠΑ. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε το κόστος παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για αυτά τα αυγά που είναι 84 ε, λεπτά του ευρώ. Το κίτρινο είναι το κόστος μεταφοράς ε, στη Γερμανία και μετά βλέπετε το κόστος που έχουμε στις υπόλοιπες χώρες. Το γαλάζιο είναι ο δασμός ε, εισαγωγής. 30,4 ευρώ στα 100 κιλά. Αυτό ήταν στο πλαίσιο του γύρου της Ουρουγουάης. Ε, βλέπετε λοιπόν ότι αυτό αποτελεί τμήμα προστασίας. Δεν έχουμε εισαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που ε, μεταπολούνται στο λιανεμπόριο. Το ίδιο ισχύει και για την ε, σκόνη του αυγού. Η διαφορά είναι ότι υπάρχει ότι ακόμα και ενώ πληρώνει η Αργεντινή τον πλήρη δασμό και πάλι είναι σε ανταγωνιστική θέση. Ζητήσαμε λοιπόν από του οικονομολόγου που συνέταξαν την έκθεση να εξετάσουν όλα τα κόστη ε, τη Ευρωπαϊκή νομοθεσία που πειράζουν τον κλάδο μας. Και τα έχουμε ε, μοιράσει σε τρει τομεί: τον περιβάλλον, την επιστημιστική ασφάλεια και τρίτον την ευημερία των ζώων, την ορθή του μεταχείριση. Αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για ε, εύλογε ανησυχίε των, Ευρωπαϊ... των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν είμαστε κατά της νομοθεσία αυτής. Εδώ βλέπετε στον κόκκινο ε, κύκλο ότι σχεδόν το 9% ε, του κόστους παραγωγής ενός κιλού αυγού στην Ευρώπη προκύπτει κατά συνέπεια της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την επιστηστική ασφάλεια, την ε, προστασία του περιβάλλοντος και την ευημερία των ζώων. Ενώ οι τρίτες χώρες δεν έχουν αντίστοιχες δαπάνες. Επομένως έχουμε ανταγωνιστικό μειονέκτημα ευθύς εξ αρχής. Να το θέσω διαφορετικά. Εάν θυμάστε, πριν από την ε, απαγόρευση των συμβατικών κλοβών στην Ευρώπη, αν είχαμε το 100 βασικό δίκτυο, όταν περάσαμε στις, στους διαθετημένους ε, κλοβούς το 2012 στην Ευρώπη, το κόστος αυξήθηκε κατά 7% για μας. Σημαντικό επίσης να επισημάνουμε ότι πολλές τρίτες χώρες ήδη ήταν ανταγωνιστικές προς εμάς, ακόμα και πριν από την απαγόρευση των, ε, κλωβών, των συμβατικών κλοβών. Και αν το περάσουμε σε άλλο επίπεδο ακόμα, βλέπετε ότι με το κόστος της οδηγίας για την ευημερία των ζώων, το κόστος για μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κόστος που προκύπτει από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ανέρχεται στο 15%. Αυτό είναι πραγματικά τεράστιο ποσοστό γιατί η παραγωγή αυγού στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να τηρήσουν τις, ε, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες και να καλύψουν και τις προσδοκίες των ε, καταναλωτών έχουν επενδύσει πάνω από 4 δις ευρώ μέχρι το 2012. Αυτό είναι πραγματικά διόλου καταφέρουν το ποσό. Βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια κάτι αντίστοιχο με την προηγούμενη. Βλέπετε ότι αν προσθέσουμε το κόστος της ε, οδηγίας ε, για την ευζοία των ε, ζώων, ανεβαίνουμε κατά 6 cent λεπτά του ευρώ ανά κιλό. Αλλά για τα αυγά δεν είναι τόσο σημαντικό, γιατί βλέπετε ότι με τον εισαγωγικό δασμό υπήρχε μια προστασία. Και όπως ξέρετε έχουμε στην Ευρώπη πολύ αυστηρή νομοθεσία για τη σαλμονέλα. Και έτσι καμία χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός Νορβηγίας και Ελβετίας δεν έχουν ε, την αδειοδότηση να εξαγάγουν ε, αυγά προς ε, την Ευρώπη για να μεταπολιθούν στο λιανεμπόριο. Ωστόσο, αυτό είναι η κατάσταση για τα αυγά με κέλυφος. Όταν περνάμε όμως στα προϊόντα αυγού, ε, η κατάσταση αλλάζει πολύ. Βλέπετε εδώ το πράσινο τμήμα που έχει ε, αυξήσει το κόστος για μας και θυμάστε που ανέφερα προηγουμένως στην Αργεντινή. Ξαφνικά βλέπετε λοιπόν ότι τα προϊόντα αυγού από την Αργεντινή, τα αποξηραμένα που έρχονται στην Ευρώπη, ακόμα και με τον πλήρη εισαγωγικό δασμό, ε, και πάλι βρίσκονται στην ίδια τιμή με αυτήν ε, στην οποία πουλάμε εμείς τα προϊόντα μας στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν πρόβλημα εδώ. Στην έκθεση ε, συμπεριλάβαμε και ορισμένα σενάρια. Όπως θυμάστε λοιπόν όταν είχαμε τις ευρωμετεύσεις της Δόχα υπήρξε ένα σχέδιο ε, εγγράφου, όπου προτινόταν ε, να υπάρξει μια μείωση κατά 50% στους εισαγωγικούς δασμούς. Είπαμε λοιπόν στους οικονομολόγους μας, ε, για να είμαστε συνεπείς με τις προηγούμενες μελέτες, ας βάλουμε την ίδια μείωση. Και να έχουμε και μία μεταβλητή ανάλογα με την ισοτιμία, τη συναλλαγματική ισοτιμία. Όμω, το πρόβλημα τώρα είναι ότι με όλες τις διμερεί διαπραγματεύσει που λαμβάνουν χώρα, πρόκειται για ελεύθερες ε, συμφωνίες, εμπορικέ συμφωνίες, που ενέχουν ε, την ε, άρση εισαγωγικών δασμών. Και για να δείτε σχηματικά, βλέπετε εδώ πώς μεταβάλλονται σχεδόν καθημερινά οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταξύ των ανταγωνιστικών προς χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πιο σημαντική διαφάνεια σήμερα το απόγευμα είναι αυτή εδώ. Δείχνει ξεκάθαρα ότι αν μειώσουμε κατά 50% τον εισαγωγικό δασμό και έχουμε και μία μεταβλητή του 10% στην συναλλαγματική σου τιμία, και εδώ μιλώ για την ε, σκόνη αυγού, όλες αυτές οι τρίτες χώρες λοιπόν ξαφνικά είναι πολύ πιο ανταγωνιστικές από εμάς. Και όπως είπα, οι διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις συνήθως ε, καταλήγουν σε, ελεύθερες, ε, σε συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Επομένως μπορείτε να βγάλετε και αυτό το γαλάζιο κομμάτι ακόμα. Τότε το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο βεβαίως. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη και συμπερασματικά, Πρόεδρε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε σχετικά μικρές διαφορές στο κόστος παραγωγής μεταξύ κρατών μελών. Αν δείτε όμω τρίτε χώρε, όπως αυτέ που ανέφερα προηγουμένως, οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Αργεντινή έχουν ένα πλεονέκτημα σε ό,τι αφορά το κόστο παραγωγής που αγγίζει το 25%. Οι εισαγωγικοί δασμοί είναι σύνομα μέσα προστασία τη Ευρωπαϊκής Βιομηχανία Αυγού και των τεράστιων επενδύσεων που έχουν πραγματοποιήσει οι ε, γεωργοί μα ε, προϊόντα αυγού. και έχουμε πολλέ νομοθετικές διατάξει για την προστασία του περιβάλλοντος, των ζώων και την επιστημική ασφάλεια. Εμείς κυρίε και κύριοι πιστεύουμε στο δίκαιο εμπόριο και όχι στο ελεύθερο εμπόριο με κάθε κόστο. Αυτό μάλιστα θέλουν και οι Ευρωπαίοι καταναλωτές. Τι θα γίνει λοιπόν στο μέλλον. Ουσιαστικά θέλουμε ένα συνδυασμό του, του αυξημένου κόστους ε, μαζί με τις ε, μειώσεις ή τις εξαλείψεις δασμών. Αυτή η κατάσταση λοιπόν θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της ανταγωνιστικής μας θέσης. Και ξέρετε ότι σε τρίτες χώρες ε, οι όρνηθες ε, ζουν κάτω από πολύ χειρότερες συνθήκες. Μάλιστα, δεν γνωρίζω καμία τρίτη χώρα που να έχει οποιαδήποτε εθνική νομοθεσία για την ευημερία των ζώων ή των ε, ονήθων σε αυτές τις χώρες που είναι βασική εμπορική εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι ζητούμε λοιπόν Πρόεδρε, τι ζητάμε από εσάς και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να ε, λάβουμε το καθεστώς του ευαίσθητου προϊόντος και να έχουμε ε, δασμολογικές γραμμές που να θεωρούνται ότι διακινδυνεύουν ότι βρίσκονται σε κίνδυνο. Έχουμε 8 τέτοιε ε, δεσμολογικέ γραμμέ. Χρειαζόμαστε επίση ε, πρότυπα ευημερία των ε, ζώων, τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε όλε τι διμερεί, αλλά και πολυμερεί ακόμα, καλό θα ήταν και στον ΠΟΕ, εμπορικέ διαπραγματεύσει. Επομένω, οτιδήποτε εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση απ' έξω θα πρέπει να πληρεί τα υψηλά μας πρότυπα ε, επιστημιστικής ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και των ζώων. Και εμείς αυτό αποκαλούμε δίκαιο εμπόριο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μακ Νομίζω ότι ήταν σημαντικές αυτές οι σκέψεις είναι θέματα που εμείς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και να αποφύγουμε στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και αδικαιολόγητες εισαγωγές από χώρες οι οποίες δεν τηρούν τα ίδια επίπεδα ασφαλείας και έχουν φυσικά πολύ χαμηλότερο κόστος από ό,τι υποχρεώνονται να έχουν η δική μας παραγωγή σε σχέση με την ποιότητα την οποία αναμένουμε. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και ελπίζω ότι με την συνεισφορά σας σήμερα θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μίκαελ Βούρτσερ της Αυστριακής Ομοσπονδίας Πουλερικών που θα μας μιλήσει για τη χρήση των συμβατικών κλοβών και για μελλοντικές προσδοκίες των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλωσορίζω τον κύριο Βούρτσερ Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Ένωση Παραγωγών Πουλερικών που εκπροσωπούνται στην αίθουσα αυτή. Έχετε κύριε Βούρτσερ το λόγο. Gentlemen. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μια πολύ θετική ευκαιρία να είμαι παρόν ενώπιον σας και να σας προσφωνήσω και να σας ομιλήσω για τα μαθήματα τα οποία έχουμε συναγάγει από την απαγόρευση στους συμβατικούς των συμβατικών κλοβών και τις προσδοκίες για τις μελλοντικές εξελίξεις από πλευράς καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας επεξηγήσω κάποιες διαφορές όσον αφορά την νομοθεσία που βρίσκουμε μεταξύ Αυστρίας και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Αυστρία απαγορεύσαμε τους συμβατικούς κλόβους ήδη τρία χρόνια πριν από τις περισσότερες χώρες μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέποντας προς το παρελθόν ήταν μια καλή απόφαση αυτή που λάβαμε πιστεύουμε. Και μπορέσαμε να συναγάγουμε νέα εμπειρία και πείρα στην αγορά και στην αγορά έχουμε περισσότερες οτόκες ε, ε, όρνηθες από ό,τι στο παρελθόν με συμβατικούς κλωβούς. Κάτι άλλο ως διαφορά είναι ότι επετράπει να δημιουργούνται εκτροφία με μικτούς κλωβούς μέχρι τα τέλη του 2004 και αυτή τη στιγμή λιγότερο από 15 εκτροφία έχουν απομείνει όπου χρησιμοποιούνται ακόμα τέτοιοι κλωβοί. Έχουμε και κάποιες διαφορές επιπλέον όσον αφορά τις διαφορετικές διατάξεις, όσον αφορά θέματα συστηματικής εκτροφής. Αλλά δεν θέλω να επισέλθω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Το ενδιαφέρον, ενδιαφέρον είναι ότι από το 2010 έχουμε ε, και ελεύθερης ε, βοσκής ε, τέτοιες οτόκες όρνηθες και τις ταΐ γεμίζουμε με ε, σόγια, το οποίο είναι σημαντική εξέλιξη. Αυτό εξοικονομεί σημαντικά κονδύλια και μπορούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να χρησιμοποιούμε αυτά τα κονδύλια και για την ίδια την αγορά. Πώς είχε η μεταβατική περίοδος σε σχέση με την αγορά, αν δούμε το λιανικό εμπόριο που είναι σίγουρα η πιο σημαντική αγορά για την, α, τους παραγωγούς της Αυστρίας. Είχαμε το νομοθέτημα ευζοίας των ζώων το 2004 στην Αυστρία. Και ήδη δύο χρόνια πιο πριν ξεκίνησαν ε, οι ε, εκτροφείς να δημιουργούν νέες μονάδες εκτροφής και ταυτόχρονα το λιανικό εμπόριο αγόραζε τα αυγά από την παραγωγή από αυτούς τους εκτροφείς απευθείας και δεν αγόραζε από τους κλοβούς. Πράγμα το οποίο ήταν πολύ θετικό για μας, γιατί διαφορετικά θα υπήρχαν πολλά προβλήματα. Και το ποσοστό α, των αναγκών μας α, επιτόπου στην Αυστρία είναι 83% της τροφοδότησής μας. Έχουν εξοικονομήσει πολλά κονδύλια οι εκτροφείς και οι ε, γεωργοί. Θα επανέλθω σε αυτό στη συνέχεια τι έγινε σε σχέση με την Αυστρία και πώς έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Έχουμε 10% περίπου οργανική παραγωγή και βλέπουμε ότι έχουμε και μεγάλο αριθμό, περίπου 19% ελεύθερης βοσκής. Έχουμε και ένα ε, ποσοστό, ε, μεγάλο ποσοστό σε συστήματα εκτροφής και ε, μονάδες εκτροφής από πλευράς αγροκτημάτων και έχουμε και διευθετημένους ε, κλόβους ε, που απομένουν ακόμα σε ένα μικρό ποσοστό στην Αυστρία. Ας δούμε τώρα τους καταναλωτές, ε, πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε τις απόψεις των καταναλωτών. Τι επιθυμούν οι καταναλωτές. Υπάρχουν διάφορες μελέτες και σφιγμομετρήσεις που έχουν γίνει και εξετάζουμε το θέμα της σπουδαιότητας των ετικετών της συσήμανση ε, όσον αφορά τα προϊόντα και τα τρόφιμα. Και όπως μπορείτε να δείτε στην ε, διαφάνεια σε σχέση με τα αυγά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα αυτά για τους καταναλωτές στην Αυστρία και θεωρείται πολύ σημαντικό να έχουν τέτοια ετικετοποίηση ή επισήμανση και βλέπετε ότι οι ετικέτες ποιότητας είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση και για τα πουλερικά πέρα από τα αυγά σε σχέση και με τα άλλα προϊόντα. Και αν πάει κανείς και επισέλθει περισσότερο στα στοιχεία αυτών που έχουν συλλεγεί και των σφιγμομετρήσεων, τι θεωρούν σημαντικό για την ποιότητα οι καταναλωτές, αν θα μπορούσε κανείς να δει πάνω-πάνω τα θέματα υγείας και της ε, ασφάλειας των τροφίμων ε, τα προϊόντα πρέπει να μην έχουν σαλμονέλα, να είναι ελεύθερα από σαλμονέλα. Είναι πολύ σημαντικό να είναι εύγευστα, να είναι, να είναι νόστιμα αυτά τα προϊόντα, να έχουν την νοστιμιά τους. Μετά αμέσως από αυτά τα κριτήρια όμως έχουμε και την περιφερειακή τοπική παραγωγή που είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους καταναλωτές και επίσης ε, η εγγύηση ευζοίας των ζώων κατά την εκτροφή. Ποια είναι η πραγματικότητα στις αγορές. Είναι σημαντικό και αυτό πολύ σημαντικό. Επικεντρωνόμενοι στην αυστριακή αγορά, τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι η Παραγωγή, παράγουν σχεδόν αποκλειστικά για το λιανικό εμπόριο. 34% αγοράζει το λιανικό εμπόριο των παραγωμένων στην Αυστρία αυγών. 22% των αυγών αγοράζονται από την μεταποιητική βιομηχανία και περίπου 40% από την γαστρονομία γενικά ως τομέα, ξενοδοχεία, μαγειρία ή άμεσες αγορές από τα εκτροφία. Και έχουμε και την παράδοση 4% περίπου των πασχαλινών αυγών, την χρήση αυτή στις οικογένειες και που στις αγορές έχει αυτή την προοπτική, μπορείτε να φανταστείτε ότι και οι τιμές έχουν σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα για τη μεταποιητική βιομηχανία και είναι <clears throat> μεγάλης σπουδαιότητας και για τον γαστρονομικό τομέα και για τα μαγειρία, τις κουζίνες κτλ. Ε, και της, ε, τη δυνατότητα επιλογής και αγοράς ακόμα και των πιο ακριβών αυστριακών τοπικών ε, περιφερειακών αυγών. Τι θέλουν οι καταναλωτές τώρα όσον αφορά την σήμανση και τις ετικέτες. Από μια άλλη μελέτη βλέπουμε ότι είναι πολύ σημαντικά τα θέματα ετικετοποίησης και συσκευασίας και σήμανσης για τους καταναλώτες. Υπάρχει μια μελέτη που λέει 86% των όσων απάντησαν σαφώς προτιμούν τοπικά περιφερειακά αυγά αυστριακής προέλευσης. 92% από όσους συμμετείχαν δεν θέλουν καθόλου αυγά από συστοιχίες κλοβών, από κλοβούς, ούτε και σε μεταποιημένα προϊόντα και θα πρέπει εδώ να υπάρχει και σαφής ε, ένδειξη στις ετικέτες ε, υπέρ των τοπικών προϊόντων, υπέρ ε, των προϊόντων ποιότητας, ποιοτικών τροφίμων και ζητούν οι καταναλωτές υποχρεωτική δεσμευτική σήμανση στην ετικετοποίηση και συσκευασία όσον αφορά και την εκτροφή και τα γαστρονομικά προϊόντα μεταποίησης. Και στη διαφάνεια τώρα μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει σε σχέση με τα διαφορά και σε σχέση με τις παραγωγές. Υπάρχουν λίγα κράτη ε, μέλη τα οποία έχουν ε, ε, πλεόνασμα σε αυτά τα αυγά. Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν έλλειμμα, είναι λιματικά σε σχέση με αυτό το προϊόν. Και γενικότερα θα ήθελα να πω ότι το σύστημα ετικετοποίηση, ενιαίας ετικετοποίηση είναι ένα τέλειο σύστημα για την Ευρώπη, λειτουργεί πολύ καλά και δίνει πολύ θετικές πληροφορίες στους καταναλωτές. Όταν έρχεται η χρονική η ώρα όμως να έχουμε μεταποιημένα προϊόντα και σε σχέση με ε, κλωβούς και δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Στην παρουσίασή μου σήμερα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε καλύτερο σύστημα ετικετοποίηση όσον αφορά την προέλευση και την εκτροφή σε σχέση με τα αυγά και αυτά τα προϊόντα. Και σχεδόν ολοκληρώνω την παρουσίασή μου και θα ήθελα να σας πω ότι αυτά που απαιτούνται σήμερα είναι να υπάρξουν δυνατότητες επενδύσεων σε σχέση με το να υπάρξει δράση στην ε, παραγωγή, την ζωική παραγωγή και να μην υπάρχει το πρόβλημα της μη αντιστοιχίας σε σχέση με τις διατάξεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλά πρέπει να γίνουν για να αποφύγουμε τέτοια προβλήματα στο μέλλον το δικό μας, το δικό μας συμπέρασμα ποιο είναι, ότι χρειαζόμαστε σαφείς πληροφορίες για τους καταναλωτές όσον αφορά τα συστήματα εκτροφής ζώων και την προέλευση των προϊόντων αυτών και θα πρέπει να είναι δεσμευτικού χαρακτήρα όχι μόνο για τα αυγά με φώσα αλλά και με τα γενικότερα προϊόντα να υπάρξει μια δικαιότερη αγορά. Γιατί? Για να είναι σεβαστές οι επιθυμίες των Ευρωπαίων καταναλωτών που θέλουν να απαγορεύονται οι κλοβοί ως τρόπος παραγωγής. Και είναι σημαντικό αυτό. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ένα δίκαιο εμπόριο και δίκαιο ανταγωνισμό για τους εκτροφείς. Και είναι αναγκαίο λοιπόν γι' αυτό να διασφαλιστούν οι πτυχές της ασφάλειας των ζώων, της, ασφα... της υγείας των ζώων και της ευσοίας των ζώων για το μέλλον. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Βούρτσελ. Τώρα θα μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τις παρουσιάσεις δίδοντας το λόγο στον κύριο Νιεβαντόφσκι. Ο συνάδελφος ο Λέινιτσακ με διορθώνει. Ο κύριος Νιεβιαντόφσκι είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φάρμιο στην Πολωνία και θα μας μιλήσει για το πώς θα οικοδομηθεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για τη βιομηχανία αυγών στην Ευρώπη μέσω της αντίληψης ε, των καταναλωτών. Οι συνάδελφοι μπορεί να δηλώσουν συμμετοχή στη συζήτηση εφόσον το επιθυμούν. Chairman. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευρωβουλευτές, Κυρίες και κύριοι, για τα επόμενα 15 λεπτά θα έχω αυτή την παρουσίαση και θα προσπαθήσω να απαντήσω στο ερώτημα πώς να δημιουργήσουμε συγκριτικά πλεονάσματα για την ε, βιομηχανία στην Ευρώπη μέσω της προσέγγισης όπως βλέπουν τα πράγματα οι καταναλωτές. Με άλλα λόγια, η προσέγγιση των καταναλωτών είναι το κρυφό όπλο, κρυφό όπλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προστατευτεί η αγορά μας από αυγά τρίτων χωρών. Για να εισαγάγω, να σας παρου, αυτοπαρουσιαστώ. Είμαι ο Ρόμπερτ Νιεβιαντόμσκι. Εκπροσωπώ την εταιρεία Φάρμιο. Είμαστε επικεφαλής ως εταιρεία στα αυγά με κέλυφο στην Πολωνία ιδρυθήκαμε και διαχειριστήκαμε την, ε, ιδρύθηκε και διαχειρίστηκε η εταιρεία μας από μια πολύ επιτυχή ομάδα εδώ και 20 χρόνια με πείρα 20 ετών. Τι είναι ενδιαφέρον ότι είμαστε επικεφαλής ως φάρμιο, ως εταιρεία και 12 μπορούμε να πούμε, ε, εδώ και 12 μήνες, από, από 12 μήνες και είναι πολύ σημαντικό αυτό το καταφέραμε με το μυστικό κρυφό μας όπλο που είναι η κοινοποίηση και επικοινωνία για τα ποιοτικά μας προϊόντα και η δουλειά που κάναμε για να ανταποκριθούμε στις απόψεις και προσεγγίσεις των καταναλωτών. Τι γνωρίζουμε για την ευρωπαϊκή βιομηχανία ότι χρειάζονται προδιαγραφές και διατάξεις για την ε, εκτροφή και την ασφάλεια και την ευζοία των ζώων. Και όλα αυτά στοιχίζουν περίπου 15%. Αυτό είναι το 15% ζήτημα το οποίο έχουμε και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως πρόβλημα έναντι των εισαγωγών προϊόντων από τρίτες χώρες. Και τώρα θα ήθελα να ρίξουμε μια ματιά στην εισαγωγή το 2012 διευθετημένων κλοβών στην αγορά της Πολωνίας. Είναι η έβδομη μεγαλύτερη παραγωγός στην Ευρώπη Πολωνία. Αν δούμε όμως τους κλοβούς, τι γίνεται με αυτούς. Η συμπίκνωση, η επικέντρωση των κλοβών είναι πάνω από 90%. Δηλαδή με άλλα λόγια τι λέει αυτό. Η πολωνική αγορά είναι μια αγορά από τις μεγαλύτερες ε, στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάνοντας λόγο για την ε, παραγωγή από κλωβούς. Ουσιαστικά δηλαδή στην εισαγωγή των διευθετημένων κλωβών ήταν πραγματικά μια πρόκληση που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Πρώτον, χρηματοοικονομική ε, αγορά, ε, χρηματοοικονομικό πρόβλημα. Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ήταν δυνατόν να διασφαλίσουν τη χρηματοδότησή τους για να προσαρμοστούν. Ήταν λοιπόν έτσι πολλοί παραγωγοί που αποσυρώντουσαν ή αποσύρθηκαν από την αγορά και αυτό οδήγησε σε μη ισόρροπες σχέσεις, σε αποσταθεροποίηση της αγοράς. Διότι σε σχέση με την παραγωγή και προσφορά είδαμε ότι οι τιμές εκτοξεύτηκαν σε ύψη σε μια χρονική συγκυρία όπου οι τιμές διπλασιάστηκαν σε σχέση με τις κανονικές τιμές που ίσχυαν. Και αυτό φυσικά προσελκύει νέες επενδύσεις διότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο για να σημειωθεί κέρδος. Έτσι λοιπόν ε, ε, με ένα νέο κύμα είχαμε μια νέα κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Λίγους μήνες μετά αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα της υπερπαραγωγής. Οι τιμές μειώθηκαν, κατακριμνίστηκαν και πολλές επιχειρήσεις καταποντίστηκαν. Τα αποτελέσματα ποια ήταν. Τα αποτελέσματα ήταν ότι έπρεπε να μειωθεί η παραγωγή από πλευράς μας. Και πράγματι ήταν μεγάλο το ζήτημα της σφαγής. Έγινε μια πολύ μεγάλη σφαγή. Και αυτό ήταν δραματική κατάσταση. Βλέποντας λοιπόν την εισαγωγή των διευθετημένων κλοβών στη χώρα μας, ήταν, μπορούμε να πούμε, μία ε, για την βιομηχανία μία τεράστια προσπάθεια. Για ποιους έγινε αυτή η τεράστια προσπάθεια. Για τους καταναλωτές, μάλιστα. Φυσικά για τους καταναλωτές. Θέλαμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και τις επιθυμίες των καταναλωτών. Τώρα το ερώτημα, το ζήτημα είναι ότι τι ακριβώς πιστεύουν και ποια είναι η άποψη των καταναλωτών γι' αυτό. Έγινε λοιπόν μια συλλογή στοιχείων δειγματοληπτικά στην πολωνική αγορά. Ζητήθηκαν οι απόψεις ε, των ε, καταναλωτών και έγινε δειγματοληπτικά από μια, μια αντιπροσωπευτική ομάδα ε, η συλλογή στοιχείων. Τι λένε οι πολίτες. Πρώτα απ' όλα λένε η ερώτηση ήταν γνωρίζετε εσείς το θέμα της ευζωίας των ζώων και το πρόγραμμα για την ευζοία των ζώων. Οι περισσότεροι από τους πελάτες, 69% είπαν όχι, δεν το γνωρίζουμε, αγνοούμε για την, την ύπαρξη αυτού του προγράμματος. 31% το γνώριζε, αλλά με ποια πηγή πληροφόρησης, κάποιες φήμες ε, που κυκλοφορούσαν κατά την περίοδο της αύξησης των τιμών το γεγονός λοιπόν ποιο είναι. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπήρξε επικοινωνία σωστή σε σχέση με τα όσα δημιουργήθηκαν υπέρ των καταναλωτών προς τους καταναλωτές. Δεν τα γνώριζαν αυτά. Πέρα από αυτά ρωτήσαμε τους Πολωνούς καταναλωτές είσαστε έτοιμοι να πληρώσετε περισσότερα χρήματα για αυγά με κέλυφος αν γνωρίζετε για ένα τέτοιο πρόγραμμα ευζοίας των ζώων. 52% απάντησαν μάλιστα είμαστε πρόθυμοι να πληρώσουμε περισσότερα. 18% είπαν δεν γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να απαντήσουμε, χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες. Συνολικά λοιπόν 70% είναι η ομάδα, η κατηγορία που πρέπει να δραστηριοποιηθεί και να κινητοποιηθεί και να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Ένα άλλο θέμα είναι η αποδεκτή τιμή. 8% είναι η αποδεκτικότητα, η αποδοχή της αύξησης τιμών από τους καταναλωτές. Έχουμε λοιπόν την εξής κατάσταση. Το πρόγραμμα ευζοίας των ζώων πιστεύουν ότι αξίζει να σημειώσει αύξηση τιμών 8% των καταναλωτών. Αν το συγκρίνουμε σε σχέση με το 15% που απαιτείται για την ευζοία των ζώων στο πρόγραμμά μας, το χάσμα, το κενό είναι πολύ μεγάλο. Έχουμε άλλα πρόσθετα επιχειρήματα. Οι προδιαγραφές για την ασφάλεια τροφίμων και η προστασία του περιβάλλοντος, η εκτροφή, το θέμα της εκτροφής των ζώων και αυτά που αναφέρθηκε προηγούμενα ότι πρέπει να αυτά τα προϊόντα να είναι ποιοτικά. Έχουμε λοιπόν μεγάλο κατάλογο επιχειρημάτων υπέρ των καταναλωτών. Έχουμε την ευκαιρία να κινητοποιήσουμε πάνω από 70% των καταναλωτών, προσφέροντας περισσότερα επιχειρήματα. Και έτσι θα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν πάνω από 8% αύξησης τιμής, 12% ίσως και 15% της τιμής και να καταφέρουμε να λύσουμε το πρόβλημα έτσι. Λοιπόν, μπορώ λοιπόν να σας πω ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών μια πολύ μεγάλη δουλειά επιτρέφει, ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα έγινε για να ε, φτάσουμε στις υψηλότερες προδιαγραφές όσον αφορά αυτά τα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έλεγα μάλιστα ότι τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγονται με τις αυστηρότερες και πιο απαιτητικέ προδιαγραφές παγκόσμια. Και τούτου λεχθέντος εξαιρετική δουλειά έχει γίνει και γίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξαιρετική δουλειά από πλευράς της βιομηχανίας. Και εμείς παράγουμε τα αυγά αυτά σύμφωνα με τις πιο αυστηρές και πιο αναβαθμισμένες ε, διατάξεις και προδιαγραφές παγκόσμια. Ένα πράγμα λείπει όμως. Κάτι ξεχάσαμε. Ξεχάσαμε να το πούμε αυτό στους καταναλωτές. Δεν τους ενημερώσαμε γι' αυτό τους καταναλωτές. Ε, θα πρέπει να είμαστε περήφανοι. Και όμως δεν τους λέμε τίποτα για αυτά τα επιτεύγματα. Δεν τους τα είπαμε, δεν τους τα κοινοποιήσαμε. Ποια είναι λοιπόν η κατάσταση. Να εισαχθεί μια επικοινωνία για να ενημερώνονται οι καταναλωτές. Πρέπει να γίνει μια συλλογή στοιχείων, να ξεκινήσει μια εκστρατεία διάχυσης, διάδοσης δεδομένων και να ξεκινήσει και η ετικέτα, το σύμβολο το οποίο θα χρησιμοποιείται στις ετικέτες για τα προϊόντα όσον αφορά τα αυγά για παράδειγμα και τα μεταποιημένα προϊόντα ως τρόφιμα. Ιδιαίτερα αυτά που είπε πριν ο προλαλής σας. Έχουμε μεγάλο ζήτημα όσον αφορά την σκόνη, τα αυγά σε σκόνη και όσον αφορά την ετικετοποίηση των ε, μεταποιημένων προϊόντων με ετικέτα που θα λέει αυτά τα προϊόντα παρήχθησαν σύμφωνα με τις πιο αυστηρές και αναβαθμισμένες ε, προδιαγραφές παγκόσμια. Έχουμε πολλές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε σχέση με την αγορά Κάποιες από αυτές αναφέρθηκαν. Αλλά αν δούμε, στρέψουμε το βλέμμα στο μέλλον, υπάρχει ακόμα και μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί από πλευράς μας στο μέλλον. Πέρυσι, ο πρώην ιδρυτής της Microsoft, ο Bill Gates, ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους παγκόσμια, στον κόσμο, άρχισε να χρηματοδοτεί μια νέα επιχείρηση που αποκαλείται Beyond Eggs, πέρα από τα αυγά. Ποια είναι η ιδέα, να παράγεται η σκόνη των αυγών χωρίς αυγά. Πώς θα παράγεται, θα παράγεται φυτικά, από φυτικά προϊόντα. Η ιδέα είναι να πωλείται στις επιχειρήσεις για να παράγεται μαγιονέζα και άλλα προϊόντα. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα τρόπο ταυτοποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων μας. Ένα τέτοιο σύμβολο, μια ετικέτα που θα λέει αυτά τα προϊόντα παρήχθησαν από αυγά. Αυτά τα παρήχθησαν από αυγά που ανταποκρίνονται στις πιο αυστηρές προδιαγραφές παγκόσμια όσον αφορά την παραγωγή τους. Αυτό θα μας βοηθούσε σε σχέση με την κατάσταση όπως έχει. Το συμπέρασμα λοιπόν ποιο είναι. Πολλά έγιναν σίγουρα. Πάρα πολλά έγιναν. Πρέπει να προστατέψουμε την αγορά με ρυθμίσεις και διατάξεις για την αγορά, ιδιαίτερα βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα, ώστε μακροπρόθεσμα σε ένα μακρύτερο χρονορίζοντα να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και να πούμε στους καταναλωτές ότι τα αυγά της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγονται με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές παγκόσμια. Ευχαριστώ. Grazie, grazie anche a Robert. Ευχαριστώ λοιπόν και τον κύριο Νιεβαντόφσκι, τους ευχαριστώ όλους για την παρουσίασή τους. Νομίζω ότι μας δώσαν πάρα πολλά στοιχεία για να θέσουμε ερωτήσεις. Ποιος ε, θα τολμήσει να ξεκινήσει ο Άγνιου μετά ο Νίκολσον. Ο Άγνιου έχει πρώτος το λόγο. Δύο από τις παρουσιάσεις τις οποίες άκουσα θέλουν να με κάνουν να αυτοκτονήσω και αναρωτιέμαι πώς και δεν το πέτυχαν ήδη οι αυστριακοί παραγωγοί. Δεν ξέρω πώς καταφέρνουν να πουλάνε τα προϊόντα τους όταν είναι υποχρεωμένοι να μην αγοράζουν ε, γενετικά τροποποιημένη ε, σόγια. 700, ε, 700 λίρες ο τόνος και με ανάγκασαν στην αρχή ε, να αγοράσω σόγια ευρωπαϊκή και εγώ αλλά μετά ευτυχώς με απάλαξαν από αυτή την υποχρέωση. Εν πάση περιπτώσει τα καταφέρνουν οι Αυστριακοί. Πάντως έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει να αυξήσετε το κόστος σας κατά 7% ουσιαστικά και τα επόμενα χρόνια θα εκτεθούν οι καταναλωτές σας σε φθηνότερα προϊόντα και εμεί θα συνεχίσουμε υποτίθεται να είμαστε ανταγωνιστικοί, κάτι το οποίο δεν θα το πετύχουμε. Δεν μιλάω μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο, μιλάω για τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία που είναι στα σύνορα με την Ουκρανία. Θα είναι τόσο εύκολο για τους Ουκρανούς να στέλνουν τα προϊόντα τους στις τρεις αυτές χώρες. Και συμφέρον είναι για αυτές τις χώρες να το κάνουν. Υπάρχει άλλος ένας τρόπος πέρα από τα τέλη βέβαια, είναι η εκπαίδευση, η ονομασία και η καταγγελία των προϊόντων που δεν είναι σε σωστό επίπεδο, αλλά αυτό είναι δύσκολο να το συνειδητοποιήσουν οι ε, καταναλωτές. Από ό,τι καταλαβαίνω από τους διαπραγματευτές, Υπάρχει δισταγμός για την ετικετοθεσία τη σωστή των προϊόντων αυτών. Παρ' όλα αυτά οι καταναλωτές πρέπει να είναι ενημερωμένοι γιατί αλλιώς θα πεθάνει η βιομηχανία των αυγών στην Ευρώπη στα πλαίσια αυτής της ύφεση. Σκοτώνοντας τη βιομηχανία μας θα δημιουργούμε μεγαλύτερη ανεργία και έχετε δίκιο που έρχεστε εδώ και το καταγγέλλετε. Πρέπει να ονοματίσουμε και να καταγγείλουμε λοιπόν τους υπεύθυνους. Είναι ένας τρόπος αυτός. Για να το πετύχουμε αυτό όμως θα πρέπει να βάλουμε τη σωστή ετικέτα στα προϊόντα και τα σούπερ μάρκετ να ξεκαθαρίσουν ότι δεν αγοράζουμε προϊόντα από αυτούς οι οποίοι δεν ετικετοθετούν σωστά. Ο Πολωνός εκπρόσωπος είπε ότι το 69% των καταναλωτών δεν έχουν ιδέα για αυτές τις ιστορίες, οπότε η βιομηχανία επιβιώνει οριακά. Θυμάμαι τη βιομηχανία του χειρίου κρέατος στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου είχαμε αλλάξει ε, την παραγωγή μας ε, με πιο ανθρώπινους εισαγωγικά όρους και τελικά αρχίσαμε να εισάγουμε κρέας ε, από χώρες οι οποίες δεν το κάναν αυτό. Λοιπόν πρέπει να έχουμε μια λογική και να μην πιεστούμε στο να πτωχεύσουμε. Ευχαριστώ κύριε Άγνιο. Ευχαριστώ για την ξεκάθαρη παρουσίασή σας. Δεν ξέρω τι είναι οι λύσεις τις οποίες προτείνετε. Εμείς ακούσαμε τέτοια προϊόντα και πριν από την ε, νομοθεσία ευημερία και ευζοίας των ζώων. Είχαμε δει ότι θα είχαμε προβλήματα σε επίπεδο χωρητικότητας και ανταγωνιστικότητας. Δεν πήραμε απαντήσεις και έχουμε τώρα τις ίδιες ανησυχίες και με τις διμερείς εμπορικές ε, ε, συμφωνίες. Ε, Πόσες, πόσα ποσότητες αυγών σε σκόνη εισάγουμε από αυτές τις αγορές. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες ποσότητες. Ακούσαμε επίσης και την Αυστρία. Είναι λίγο απομονωμένη η θέση σας. Τα κέικ και τα γλυκά σας τα φτιάχνετε με αυστριακά αυγά γιατί η, τα αυγά σε σκόνη είναι ένα προϊόν θα έλεγα διεθνές και δεν έχει κάποια χαρακτηριστικά τοπικά και δεν υπάρχουν ετικέτες σε τέτοιου είδους προϊόντα για το είδος της, το, το, το, των αυγών σε σκόνη τα οποία χρησιμοποιούνται. Θα ήθελα λοιπόν να μας πει η βιομηχανία τι λύση μπορεί να βρει παρά να δίνει ε, μάχη στα πλαίσια των διμερών συμφωνιών. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα προς συζήτηση, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που κάποιοι τομείς προβλημάτων θα ξεχαστούν και φοβάμαι ότι ο δικός σας τομέας κινδυνεύει. Εμείς κάνουμε λοιπόν όλα αυτά τα σχόλια τα οποία ακούσαμε στην Επιτροπή δεν μπορούμε εμείς να πάρουμε μέρος απευθείας στις διμερείς διαπραγματεύσεις που από ό,τι φαίνεται θα βλάψουν τον τομέα σας. Θα θέλαμε όμως να μάθουμε πώς μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε. Είμαστε, ε, δυσφορούμε για την κατάσταση, αλλά στα πλαίσια των δημερών συμφωνιών θα πρέπει να προσέξετε για να μην σας αγνοήσουν και μετά θα έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία και θα είναι πολύ αργά πια για να διορθώσουμε το οτιδήποτε. Ευχαριστώ. Ο Νίκολσον έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αρχικά θα ήθελα να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία και να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα στο Κοινοβούλιο. Τουλάχιστον ε, να γνωρίζουμε κάτι που μέχρι τώρα θεωρεί το μη σημαντικό πρόβλημα, αλλά μετά τα όσα ακούσουμε από τους ομιλητές, καθίσταται σαφές ότι είναι ένα μακροπρόθεσμο σοβαρό πρόβλημα. Όπω αναφέρθηκε προηγουμένω και εμά είναι κάτι το οποίο μα προβληματίζει και μα αγανακτεί, όπω και εσά ε, σε αυτόν τον βιομηχανικό κλάδο. Ο κύριο Βόκαρ αναφέρθηκε στον τομέα των πουλερικών. Και πράγματι ήταν πολύ ελαφρύ το καθεστώς, ε, ήπιο το καθεστώς ε, στο πλαίσιο της κοινή γεωργικής πολιτικής. Βεβαίως ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι νομοθετικές διατάξεις για την ευημερία των ζώων και όλες αυτές οι αλλαγές είχαν σημαντικό αντίκτυπο σε αυτή την βιομηχανία. Και το αναφέρατε. Όμως ποιο είναι το πραγματικό κόστος. Γιατί πρέπει να αλλάξουμε δραματικά από την προηγούμενη κατάσταση και πλέον βλέπουμε ότι έχουμε φύγει από τους συμβατικούς κλωβούς Υποτίθεται ότι σε όλα τα κράτη-μέλη παράγονται με αναλεκτικές μεθόδους. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο αυτό ισχύει και αν είναι θετικό ή όχι. Από τα σημαντικά, λοιπόν, από τα συμβατικούς κλωβούς πήγαμε ε, ε, στους διαθετημένους. Κάτι το άλλο το οποίο αναφέρθηκε, νομίζω ότι ήταν ο Πολωνός συνάδελφος που το ανέφερε. 12 έως 18% πάνω ή μπορεί το ποσό να προέρχεται από τον καταναλωτή. Έχει τη δυνατότητα αυτή ο καταναλωτής σε αυτή την περίοδο. Μετά από όλη αυτή την ε, περίοδο οικονομικών δυσκολιών, για να το πω ήπια, οι καταναλωτές ε, νομίζω ότι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Και αν αυξήσουμε και την τιμή του τελικού προϊόντος ε, στο τρόφιμο που πρέπει να αγοράσουν, ουσιαστικά τους δυσκολεύουμε ακόμα περισσότερο και ίσως θα πρέπει να βρουν εναλλακτικέ για αυτό το τρόφιμο. Αυτά είναι τα προβλήματα που εντοπίζω εγώ, γι' αυτό και επανέρχομαι στο πρώτο μου σχόλιο, ότι και εμείς ε, προβληματιζόμαστε εξίσου με πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον, συμμερίζομαι όμως ε, αυτή την ανησυχία. Και νομίζω ότι είναι αυτοκαταστροφικές αυτές οι τάσεις που δείχνουμε, γιατί δεν αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα. Ότι δεν θα έχουμε τη δυνατότητα και ή θα εισάγουμε προϊόντα από αλλού αντί να, παράγουμε, να καταναλώνουμε αυτά που παράγουμε εμείς. Ξέρω ότι ο Μάρτεν δεν συμφωνεί με όλα όσα είπαμε, αλλά ε, έτσι κι θα διαφωνούμε πλήρως ε, σε αυτές τις εκλογές. Αλλά όπως και να έχει όλα αυτά γίνονται σε φιλικό πλαίσιο. Κάτι άλλο το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως. για το μέλλον της Γεωργίας. Αν δείτε οι ε, ΙΠΑ και έχουν ένα ε, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της τάξης του 25%. Αυτό είναι τεράστιο. Καθορίζει ολόκληρη την αγορά. Πώς θα γίνει αυτό λοιπόν στο πλαίσιο της, ε, των διαπραγματεύσεων TTIP, της ε, ε, εταιρικής σχέσης, το συζητήσαμε και χθες θα γίνει στους επόμενους 24-36 μήνες αυτές τις διαπραγματεύσεις. Εσείς λοιπόν σε αυτό το χρονικό πλαίσιο πώς θα ε, χειριστείτε αυτή την κατάσταση και πώς θα προσπαθήσετε να μεταφέρετε και το δικό σας μήνυμα. Γιατί θα υπάρχει ανταγωνισμός και ξέρουμε όλοι τι σημαίνουν οι διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ. Κάποιες φορές ε, είναι και ιδιαίτερα πιεστικοί. Για να μην είμαι και μόνο αρνητικός, ε, να πω για κάτι θετικό. Μπορείτε να μας πείτε για κάτι θετικό το οποίο μπορεί να γίνει μέσα στο επόμενο διάστημα για τον ε, κλάδο αυτό. Γιατί πολλοί γεωργοί ε, κατηγορούνται ότι είναι πολύ αρνητικοί και απεσιόδοξοι και όλο γκρινιάζουν. Επομένως καλό είναι να ακούσουμε και κάτι καλό. Ευχαριστώ. Thanks, Jim. Ευχαριστώ. Ρούμπιξ και μετά Κόστιγκερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ άκουσα και τις τρεις παρουσιάσεις ε, με μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες ε, και οι τρεις εκθέσεις. Όμως, από ό,τι κατάλαβα δεν ε, συμφωνούν μεταξύ τους. Εάν πούμε ότι το 70% όλων των εισαγωγών αυγού προς την Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχονται από τρεις χώρες, ΗΠΑ, Αργεντινή και Ινδία, δεν μπορούμε σε αυτή την περίπτωση να ελέγξουμε, να περιορίσουμε, να έχουμε κάποιες ε, συμφωνίες ε, επ' αυτού, να ελέγξουμε τις συνθήκες ε, διαβίωσης αυτών των ζώων και αν δεν έχουμε πληροφορίες ε, για την εκτροφή των πτηνών σε τρεις χώρες και αν δεν έχουμε αρνητική επίπτωση, ε, τότε ίσως μπορεί να οδηγηθούμε σε ένα διέξοδο. Να ανησυχούμε για την ευημερία των ζώων περισσότερο από τα ίδια τα ζώα όταν ε, κάναμε ολόκληρο αυτό το καθεστώς ήταν να έχουμε καλές συνθήκες διαβίωσης για τα πτηνά για να ε, έχουμε και καλύτερη παραγωγή. Εάν αυτό όμως δεν συμβαίνει, αν δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις ε, ζωοτροφές για τα πτηνά, τότε δεν μπορούμε να έχουμε καμία συμφωνία με αυτές τις τρίτες χώρες. Αλλά ούτε αυτό μπορούμε να το κάνουμε γιατί δεν χρειαζόμαστε τα αυγά. Τι κάνουμε λοιπόν. Μπορούμε να ελέγξουμε, να επισκεφθούμε τις τρίτες χώρες, να δούμε ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσης των ε, πουλερικών. Και σε ποιο βαθμό κιόλα να τα εξετάσουμε. Μα απασχολεί μόνο η ευημερία ε, τη όρνηθα, εντάξει. Αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Στη χώρα μου, για παράδειγμα, στη Λετωνία, έχουμε τα αυγά ποιότητα Α και Β στα καταστήματα όχι όμως επειδή έχουν ε, μεγαλύτερο κρόκο ή επειδή έχουν ε, μεταλλαγμένα ή όχι, είναι ε, ανάλογα με το μέγεθός τους. Κάποια είναι μεγαλύτερα και αυτό αναφέρεται και ότι είναι καλύτερης ποιότητας. Τώρα τι ποιότητα είναι αυτή, τι εννοούμε με τη λέξη ποιότητα, δεν το ξέρει κανείς. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και εμείς οι πολιτικοί και οι επιστήμονες. Όλοι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε γιατί πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Και αν προχωρήσουμε σε αυτή την ε, ψηφοφορία, συγγνώμη, σε αυτό το δρόμο, και διαμορφώσουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τα πουλερικά από ό,τι για τους ανθρώπους, τότε οι ε, πολίτες μας θα φύγουν από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να ανησυχούμε ότι εισάγουμε προϊόντα. Η Ελίζαμπεθ έχει το λόγο. Σε ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ τους ε, πραγματογνώμονες, τους εμπειρογνώμονες για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση που μας έκαναν τις παρεμβάσεις τους ε, για να αφυπνιστούμε ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει και ποια πίεση υφίσταται ο συνολικός τομέας στην Ευρώπη. Φυσικά με εθνικές ε, ιδιομορφίες και χαρακτηριστικά που αρκετές φορές αναφέρθηκε και η Αυστρία ήδη σήμερα επανειλημμένα. Και πιστεύω ότι κυρίως, μια και είμαστε μικρή χώρα, μια ευρύτερη στρατηγική ε, σχεδιάστηκε από την αρχή, ώστε να υπάρξει και επικοινωνία με τους καταναλωτές, γυναίκες και άνδρες, για να δοθεί η πρέπουσα ιδέουσα αξία σε αυτή την προσπάθεια και να θέσουμε και ιδιαίτερο βάρος στην ποιότητα, ποιοτικά προϊόντα Σπάνια υπάρχει τέτοια ευκαιρία να ορθοποδήσει κανεί την παραγωγή με τέτοια εγχειρήματα και πρέπει να αναζητηθούν νέες εναλλακτικέ οδοί και δυνατότητε. Και όλοι συμφωνούν γι' αυτό, το ότι η κατάσταση γενικά είναι πολύ δυσχερή, πολύ δύσκολη και φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στην αγορά. Και κάποια αριθμητικά μεγέθη, κάποιοι αριθμοί με συγκλώνησαν, ιδιαίτερα όταν βλέπουμε τι δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις διάφορες παραγωγές, ε, ε, σε διάφορους τρόπους παραγωγής και πόσα εισάγονται από αυτά τα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να υπάρξει ετικετοποίηση και επισήμανση, σήμανση, ώστε να γνωρίζουν οι, παραγωγοί, οι καταναλωτές τι προϊόντα αγοράζουν και σε ποιες προδιαγραφές ανταποκρίνονται. Τίθεται το ερώτημα σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δραστηριοποιηθεί και θέλει και πρέπει να δραστηριοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα στην ευρωπαϊκή αγορά ώστε αυτός ο τομέας να ενισχυθεί και η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα να βελτιωθεί και να ενδυναμωθεί. Δεν είναι δυνατόν και να το δεχόμαστε και το βλέπουμε. Υπάρχει διαρκώς ε, το θέμα των διμερών συμφωνιών. Δεν μπορούμε με τέτοιες διμερείς συμφωνίες να ζούμε με μόνιμο τρόπο. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει και σε σχέση με τις εξαγωγές αυτών των προϊόντων. Και ήδη προαναφέρθηκε αυτό αν θέλουμε να δούμε τι γίνεται σε, αυτήν την, σε αυτόν τον τομέα παγκόσμια, αν δεν κάνουμε κάτι, τότε δεν έχουμε ευκαιρία ως Ευρώπη να ορθοποδήσουμε και να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων στην παραγωγή. Καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει. Είναι δυνατόν να γίνουν επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα βοηθούν τις εταιρείες και θα δίνουν τη δυνατότητα τι, να παράγουν στο εξωτερικό οι βιομηχανίες μας και να υπάρχουν εκεί μονάδες εκτροφής που να μην ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά τα προϊόντα να εισάγονται πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις δικές μας αγορές και να υπονομεύουν και να καταστρέφουν τις αγορές μας. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, λάβει, να τοποθετηθεί ξεκάθαρα σε αυτόν τον τομέα. Διότι αυτός ο τομέας για τους πολίτες μας είναι πολύ σημαντικός και πρέπει κάτι να κάνουμε. Στο τέλος τέλος πρόκειται για κονδύλια φορολογουμένων πρέπει κάτι να κάνουμε ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη προώθηση, προαγωγή αυτού του τομέα. Θα ευχαριστιόμουν αν η Επιτροπή απαντούσε αυτά τα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Ο τελευταίος ομιλητής για... Σας ευχαριστώ και εγώ Πρόεδρε. Σχεδόν θυμάται κανείς τα φοιτητικά του χρόνια με όλα αυτά. Τότε όταν είμαστε φοιτητές με τα θέματα της ευζοίας των ζώων κατεβαίναμε στο δρόμο και λέγαμε να κατα... οι συστοιχίες κλοβών. Το πρόβλημα λοιπόν είναι τι γίνεται σε σχέση με τα θέματα εκτροφής ζώων και όταν έχουμε για παράδειγμα ε, την εκτροφή ε, αγελάδων για την γαλακτοπαραγωγή ή την έχουμε, όταν έχουμε την ε, εκτροφή χείρων πρέπει να έχουμε καλύτερη ευζοία ζώων και να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη αυτό το θέμα. Τώρα μεγάλωσα και ορίμασα πια και ε, ε, έχοντας δει τη σοσιαλιστική Γερμανία, την λαϊκή δημοκρατία της Γερμανίας που ήταν η πιο αρνητική πτυχή ε, που είχε στην παραγωγή αυτή και έλεγαν ότι αυτό θα ήταν το πιο ε, υγιεινό αυγό γιατί ε, τότε οι όρνηθες με, λέει, με τα πιο υγιεινά προϊόντα ως τρόφιμα και όταν ε, είχαμε κάποια θέματα ασθένειας ε, μπορούσαν αυτά μέσα σε ένα κλωβό να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα. Όταν τρέχουν ελεύθερα όμως ε, αυτά τα ζώα είναι πιο δύσκολη η αντιμετώπιση. Όμως παρόλα αυτά θέλουμε βελτιώσει στην ευζοία των ζώων. Είναι αυτονόητο αυτό όμως κάτι πρέπει να συναγάγουμε ως συμπέρασμα από όλα αυτά. Και πρέπει να πω ότι αν με τους όρους εκτροφής ζώων το κόστος της παραγωγής μας αυξάνεται, ε, τότε μόνο δύο δυνατότητες υπάρχουν. Και, και, πάντα στην Ευρώπη μιλώ τώρα, να γίνεται αυτό στην Ευρώπη, εκτροφή ζώων στην Ευρώπη και παραγωγή στην Ευρώπη. Αλλά να μην υπάρχει και ε, διαστρέβλωση ανταγωνισμού. Στην παγκόσμια αγορά όμως τι γίνεται. Κάνουν άλλα, άλλες πρακτικές ακολουθούν από ότι εμείς. Και όταν είμαστε πιο ακριβείς στην παραγωγή εμείς από ότι οι ανταγωνιστές μας στη διεθνή, στην παγκόσμια αγορά, τι κάνουμε. Πρώτη δυνατότητα. Επικοινωνία με τους καταναλωτές και ε, ενημέρωσή τους, διαφώτισή τους ότι πρέπει να υπάρχουν υψηλές προδιαγραφές και όλα αυτά κοστίζουν. Λοιπόν, σε σχέση με τη Γερμανία, ο Γερμανός όταν τρώει το πρωινό του αυγό, λοιπόν, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, θέλει να ξέρει από πού προέρχεται αυτό το αυγό και προσπαθεί να δει από, ε, η προέλευση ποια είναι και πώς έχει παραχθεί. Όταν όμως βλέπουμε τις μελέτες και αναφέρθηκε αυτό και από προλαλήσαντα, όταν έχουμε τα μπισκότα, τα κέκα, τα μεταποιημένα προϊόντα όπου χρησιμοποιούνται τέτοια αυγά, πρέπει να ξέρουμε Ποιου είδους αυγά με ποια προέλευση χρησιμοποιούνται σε αυτή τη μεταποίηση. Δηλαδή ουσιαστικά ο, παρα, ο ε, παραγωγός, ο καταναλωτής ε, σε τέτοιου είδους προϊόντα δεν μπορεί να παρακολουθήσει την αλυσίδα. Ε, πώς παράγονται αυτά και όταν ε, πρέπει κάτι να ε, πληρώνεται σε σχέση με την, ε, με, την τιμή αυτό, αυτών των προϊόντων, τότε οι καταναλωτές πολλές φορές φέρονται και διαφορετικά από ότι για το πρωινό αυγό που τρώνε στο πρωινό τους και είναι πρόθυμοι να πληρώσουν κάτι παραπάνω γι' αυτό. για θέλουν να πληρώνουν κάτι λιγότερο σε σχέση με τα, με τα ποιημένα προϊόντα. Τι θα γίνει λοιπόν, αν είμαστε πιο ακριβείς στην παραγωγή θα εξαφανιστούν τα προϊόντα μας. Δεν θα είναι δυνατόν να υποστούμε και να αντέξουμε τον ανταγωνισμό. Και φτάνουμε κάνουμε στο πρόβλημα της ενίσχυσης των ενισχύσεων και επιδοτήσεων. Τι θα κάνουμε. Κοντός ψαλμός αλληλούια. Την εντατικότητα, το βάθος ε, α, της κατάσ... των μέτρων στην Ευρώπη για την ευζοία των ζώων πρέπει να δούμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε την ευζοία των ζώων με προσιτές τιμές προϊόντων και παραγωγής. Διαφορετικά δεν θα μπορούμε να παράγουμε και πρέπει να ποσοστοποιήσουμε αναόρνηθα ή ανααυγό πόσο μεγάλο είναι το ποσοστό του πλεονεκτήματος, ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που έχουν ε, οι παραγωγοί σε σχέση με την τιμή του τελικού προϊόντος. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα μιλήσουν οι τρεις ε, ομιλητές οι οποίοι θα απαντήσουν στις ερωτήσεις. Έχουμε κάποιο εκπρόσωπο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, δεν έχουμε κάποιον. Οπότε δίνω το λόγο... Α, υπάρχει κάποιος. Εδώ είναι, δεν σας είδα. Γεια σας. Θα ήθελα να ε, μιλήσω λίγο για το πλαίσιο των παρουσιάσεων οι οποίες δόθηκαν σχετικά με την αγορά των αυγών. Να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγει ε, περισσότερα από ό,τι περιορίζει, από ό,τι εισάγει. Νομίζω ότι είναι πολύ περιορισμένες οι εισαγωγές και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Δεύτερον, σε μία από τις παρουσιάσεις άκουσα ότι το 17% της αγοράς αντιπροσωπεύεται από ολόκληρα αυγά, αυγά με κέλυφος. Και η αγορά αυτή είναι αρκετά προστατευμένη, έχουμε πολλά υψηλά επίπεδα προστασίας και υπάρχουν ελάχιστες τρίτες χώρες οι οποίες ε, μπορούν να εξάγουν αυγά με κέλυφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Για τα προϊόντα αυγών έχουμε το 30% που καλύπτεται από εισαγωγές. Καταλαβαίνουμε βέβαια στις παρουσιάσεις που έγιναν ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές στο κόστος παραγωγής. Αυτό οφείλεται εν μέρη και στους κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ευημερία των ζώων, τις απαιτήσει για τις ζωοτροφές κτλ. Ακούστηκε και από έναν από τους ομιλητές επίσης ότι είναι και κάτι το οποίο μας επιτρέπει να έχουμε μια σωστή αγορά στον τομέα των αυγών. γύρω από τις διαπραγματεύσεις τις εμπορικές και τις διμερείς κυρίως διαπραγματεύσεις. Να υπογραμμίσω εδώ ότι στην περίπτωση των διαπραγματεύσεων αυτών έχουμε να κάνουμε με ένα πακέτο στο σύνολό του όπου καλύπτονται πάρα πολλά προϊόντα και εμείς προσπαθούμε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης να καλύψουμε το σύνολο των νομοθετικών ρυθμίσεων στα πλαίσια αυτών των διαπραγματεύσεων. Προσπαθήσαμε να εισάγουμε ιδέες και νομοθετικά επίπεδα προστασίας στον τομέα ιδιαίτερα της ευζοίας. Τι άλλο θα ήθελα να προσθέσω. Ακούστηκαν ορισμένα πράγματα για την ποιότητα. Εμείς έχουμε υψηλά ποιοτικά επίπεδα και για την εμπορία των αυγών με κέλυφος ε, και για τη σωστή ετικετοθεσία, ειδικά για τα αυγά και έχουμε επίσης και ένα πάρα πολύ καλό σύστημα ίχνηλασιμότητας της προέλευσης και του συστήματος εκτροφής. Όταν δηλαδή αγοράζει αυγά ο καταναλωτής μπορεί όλα αυτά να τα μάθει. Αυτά έχουμε κάνει για τον τομέα. Έχουμε θετικές ανταποκρίσεις σχετικά με την ασφάλεια του τροφίμου αυτού και των μέτρων ασφαλείας που λαμβάνονται για την παραγωγή ολόκληρων αυγών. Για τα υποπροϊόντα αυγού ακούστηκε πάρα πολύ συχνά ότι διάφορα τμήματα των παραγωγών θέλουν να υπάρχει εκεί αναφορά και στην προέλευση και την ποιότητα των προϊόντων αυγού. Γίνεται μια μελέτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα επεξεργασμένα τρόφιμα και στόχος αυτής της συγκεκριμένης έρευνας θα είναι η προετοιμασία μιας έκθεσης για τον τρόπο με τον οποίο τα τρόφιμα στα τρόφιμα θα υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης ε, ενός προϊόντος ιδιαίτερα όταν ξεπερνάει το 50% του περιεχομένου. Εμείς θα παρουσιάσουμε και στο Συμβούλιο και σε εσά το αποτέλεσμα της έρευνας και της μελέτης και τις διάφορες επιλογές. Θα συμπεριλάβουμε στην έρευνα αυτή και τα προϊόντα αυγού. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί και θα δούμε τι δράση μπορούμε να αναλάβουμε από εκεί και πέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Βουίλιαμς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και για τα ερωτήματά σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσα μπορώ περισσότερα. Κύριε Μαγκίνες, ρωτήσατε τι ποσοστό ή τι ποσότητες ε, σκόνης ε, αυγού εισάγουμε από το εξωτερικό. Αν δείτε ότι, ε, ότι υπάρχει ένα κόστος της μεταφοράς του νερού που εμπεριέχεται μέσα σε ένα αυγό, ε, είναι καλύτερο να ε, μεταφερθεί αφιδατωμένο το προϊόν. Οι εισαγωγές που έχουμε λοιπόν στις, ε, στη σκόνη κρόκου, γιατί είμαστε καθαροί καταναλωτές αυτού του προϊόντος, τότε βλέπουμε ότι τα περισσότερα προϊόντα που εισάγουμε από κάποιες χώρες εκτός Ελβετίας, γιατί πράγματι και, αυτές, και από αυτή τη χώρα εισάγουμε, σε μεγάλο ποσοστό λοιπόν πρόκειται για αποξηραμένα τρόφιμα. Μετά, ερώτημα του κυρίου Νίκολσον. Πώς θα διαχειριστούμε αυτό το 25% το μειονέκτημα που αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να σας πω, εκπροσωπώντας και τους ε, παραγωγούς, ότι απέχουμε πολύ από την ε, ιδανική κατάσταση. Βεβαίω και ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, σκαμπανεβάσματα στην αγορά, αλλά ουσιαστικά μας ε, καλούν να βελτιώσουμε, να αλλάξουμε άρδιν και να βελτιώσουμε σε πολύ σημαντικό βαθμό τον τρόπο παραγωγής μας. Το κάναμε αυτό, αλλά δεν ζητούν κάτι αντίστοιχο από τις τρίτες χώρες. Εμά δεν μας απασχολεί τι πρότυπα ε, τηρούν στις δυτικέ τους χώρες, αλλά αν θέλουν να εξαγάγουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα πρέπει να πληρούν τα ίδια πρότυπα με εμά. Γιατί ιδάλλως οδηγούμεθα σε αυτό το μειονέκτημα το 25%, το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η προστασία από του ε, εισαγωγικού δασμού που είναι και εύλογο να υπάρχουν. Τρίτο σημείο. Όπως είπε και η κυρία Πανεφάς από την Επιτροπή, πράγματι δεν εισάγουμε τεράστιες ποσότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτω από το 1% της ευρωπαϊκής ε, κατανάλωσης ε, εισάγεται και εμείς εξάγουμε περίπου 3,5% από την ευρωπαϊκή παραγωγή. Επομένως υπάρχει αυτάρκεια. Όμως εμείς ε, έχουμε το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον και εκεί με τις διάφορες συμφωνίες που θα υπάρξουν θα τεθούμε εκτός της διεθνούς αγοράς εξαιτία του κόστους και θα επιτρέψουμε και εισαγωγέ στην Ευρωπαϊκή, μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εισαγωγέ που είναι πιο ανταγωνιστικές από τα δικά μας προϊόντα. Είμαι ρεαλιστής, ε, ξέρω ότι οι τιμές των ζωοτροφών είναι πιο φτηνέ ε, στη Λατινική Αμερική, χώρες όπως ε, η Αργεντινή έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα όμως δεν έχουν την ομοθεσία την οποία εμείς θα πρέπει να τηρούμε. Γι' αυτό επανέρχομαι στο σημείο προβληματισμού που ανέφερα προηγουμένως. Κάτι άλλο το οποίο αναφέρθηκε είναι ότι η Επιτροπή προσπάθησε να εντάξει την ευημερία των ζώων στις διμερείς διαπραγματεύσεις. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε στη συμφωνία που τελικά δεν υπεγράφει με την, Ουκρανία. Εάν είχε υπογραφεί αυτή η συμφωνία, τότε όταν θα είχαν ε, χειριστεί το πρόγραμμά τους ε, για την ε, προστασία από τη σαλμονέλα, τότε θα είχαμε περάσει σε άλλη κατάσταση σε ό,τι φορά την εισαγωγή αυγών. Ξέρετε βέβαια ότι δεν υπεγράφει συμφωνία, επομένω έχει μετατεθεί για κάποια στιγμή στο μέλλον. Εγώ επισκέφθηκα την Αργεντινή πριν από 2-3 χρόνια και πήγαμε σε μία επιχείρηση που ήθελε να εξαγάγει προς την Ευρώπη. Ο ιδιοκτήτης μα είπε πολύ ρεαλιστικά, ξέρω ότι αν θέλω να εξαγάγω προς την αγορά σα στην Ευρώπη, πρέπει να τηρήσω τα πρότυπά σας. Όχι ότι είμαι αναγκασμένο από την νομοθεσία, αλλά επειδή οι καταναλωτές που θα αγοράσουν τα προϊόντα μου στην Ευρώπη απαιτούν να τηρήσω τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Επομένως, ε, Βλέπουμε ότι η αγορά θα επιβάλλει τα πρότυπά της ε, στο μέλλον, όμως και πάλι χρειαζόμαστε κατά βάση οι επιχειρήσεις, και οι επιχειρήσεις που θέλουν να εξαγάγουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να γνωρίζουν ξεκάθαρα και εκ των προτέρων ότι θα πρέπει να πληρώσουν κάποια κριτήρια. Και τέλος, ε, η κατάλληλη σήμανση για την ετικετοθεσία πάνω σε κάθε αυγό είναι πραγματικά μια καταπληκτική ιδέα. Το πρόβλημα είναι ότι όταν βγάζουμε το αυγό από το κέλυφος, τότε τα πράγματα μπερδεύονται πολύ εύκολα και γρήγορα. Και οποιαδήποτε μορφή δικαιοθεσίας ε, προς ενημέρωση των ε, καταναλωτών μας, των πελατών, που μπορεί να είναι και ο κλάδος της μεταποίησης, θα βοηθήσει. Σίγουρα και συνάδελφοι θα έχουν κάτι να προσθέσουν, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μάρκ. Ο Μίκαελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Πολλά έχουν ήδη απαντηθεί από τον το Μάρκ. Ερώτηση. Ποιος πληρώνει το υψηλότερο ε, ποσό ως τιμή για αυτό το προϊόν στην Αυστρία. Οι καταναλωτέ που αγοράζουν τα νοπά φρέσκα προϊόντα πληρώνουν αυτά τα, αυτές τις υψηλότερες τιμές. Έχετε σίγουρα δίκιο όμως όταν λέτε, λέτε ότι είναι δύσκολο να πουλάμε προϊόντα με τόσο υψηλή διαφορά τιμής και να μπορούν ε, να αντιμετωπίζουν ευρύτερα αυτό το θέμα η παραγωγή. Ρωτήθηκε ποιο είναι το ποσοστό μεταποιημένων ε, τέτοιων ε, ε, στη μεταποίηση τέτοιων, τέτοιων προϊόντων σε σχέση για παράδειγμα με τα ζυμαρικά ή άλλα είναι λιγότερο από 10% αλλά μάλλον επειδή δεν υπάρχει κάποια σήμα, επισήμαση, ετικετοποίηση και αναφορά απουσιάζει αυτή η πληροφορία για τους καταναλωτές και πρέπει οι καταναλωτές να παίρνουν αυτή την ενημέρωση τότε μπορεί να αλλάξει η κατάσταση στην Αυστρία έχουμε 83% αυτοτροφοδοτούμενη αγορά. Καλύπτουμε εμείς τις ανάγκες μας, έχουμε επάρκεια 83%. Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό που είπε πιο πριν ο Ρόμπερ. Πρέπει να δούμε τις ανάγκες των καταναλωτών και τις προσδοκίες των καταναλωτών. Απαγορεύσαμε τις συμβατικές ε, συστοιχίες κλοβών, τους συμβατικούς κλοβού, επειδή το ζήτησαν οι καταναλωτές. Και η παραγωγή στην Ευρώπη πρέπει να μεριμνήσουμε μακροπρόθεσμα να μπορεί να επιβιώσει. Και πρέπει να διασφαλίσουμε τις προδιαγραφές για την ε, ασφάλεια και υγεία των τροφίμων και τις προδιαγραφές για την ε, αναγκαία αυτή παραγωγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Βούτσερ. Τελευταίος ο κύριος Νιεβαντόφσκι. Ρόμπερτ, έχει το λόγο. Όχι. Μία τελευταία παρατήρηση. Ακούστηκαν πολλά. Σχετικά με την ετικετοθεσία, την σήμανση η οποία μπορεί να δείχνει την ποιότητα εφόσον πουλάμε. Αυτό δεν αφορά ο, όλες τις, όλους τους καταναλωτές. Είδατε ότι ε, οι καταναλωτές 70% είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν επιπλέον, αλλά όχι όλοι βέβαια. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να κάνουμε δύο πράγματα μαζί. Από τη μία να επιδείξουμε την ποιότητα των προϊόντων μας στις ετικέτες και στις συσκευασίες και ταυτόχρονα ε, να φροντίσουμε να έχουμε τις σωστές εμπορικές ρυθμίσεις. Γιατί η βιομηχανία μας έχει κάνει πολλές επενδύσεις, έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες και υπάρχει μια έλλειψη ισορροπίας ανάμεσα σε αυτά τα οποία έχει κάνει η βιομηχανία και στο μέγεθος της επένδυσης δηλαδή από τη μία και από την άλλη σε ποιο βαθμό οι καταναλωτές αναγνωρίζουν την επένδυση αυτή. Αυτή η απόσταση πρέπει να καλυφθεί. Και γι' αυτό λοιπόν εγώ προτείνω να ενημερώνουμε σωστά και να εκπαιδεύουμε σωστά τους καταναλωτές, κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει και εμάς, αν και αυτό βέβαια δεν είναι η μοναδική λύση στο πρόβλημα. Σας ευχαριστώ όλους και τους τρεις. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που πήραν μέρος στη συζήτηση. Τελειώνει εδώ η συνεδρίασή μας μετά από αυτήν την σημαντική συζήτηση. Υπενθυμίζω τις επόμενες συναντήσεις, συνεδριάσεις, 17η Μαρτίου και 18 από τις 3 ε, μέχρι τις 6.30. 18 Μαρτίου. Θα δούμε αν μπορούμε να ξεκινήσουμε σαν συντονιστές τώρα, αλλιώς θα ξεκινήσουμε στις 5.